Uh, Καλημέρα σε όλους. Για όσους δεν έχω δει ακόμα, καλή χρονιά. Νομίζω σας είδα στο Σασβούργο Λοιπόν, θα περάσουμε στις ψηφοφορίες σήμερα. Στις 11 θα έρθει και η Ρουμανική Προεδρία. Κάποιες ψηφοφορίες όμως ακυρώθηκαν. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μας πάρει τόσο χρόνο. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 11 λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό ε, Πρόγραμμα Σωμάτων Αλληλεγγύης. Ε, κυρία Θεοχάρη, θέλετε να πείτε κάτι πριν ξεκινήσουμε. Ήθελα απλώ να ευχαριστήσω τον Κρίστιαν και τον Χάρη για την ε, πολύ καλή δουλειά τους Τη σκληρή δουλειά του. Τη χάρη, συγγνώμη. Ευχαριστώ να ξεκινήσουμε με ψηφοφορία λοιπόν. Θα κάνουμε ένα τεστ όμως. Πρέπει να δούμε αν λειτουργούν ε, τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμαστικό είναι αυτό έτσι. Ψήφισαν 19. Πέρασε ψηφοφορία. Εντάξει μια χαρά λειτουργεί το σύστημα. Η τεχνολογία είναι μαζί μας. 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27, 28 και 100 από κοινού υπέρ κατά Α, συγγνώμη. Να τα κάνουμε ξεχωριστά. Μάλιστα, εντάξει. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104. Α, συγγνώμη. 4 έως 31 Μποκινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ 107 άρχιτη ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 11 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 να το ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία το 111. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 100... 113. Όχι, συγγνώμη, 112. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε το 116 παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 12-8 θέλουμε να ελέγξουμε κάτι σχετικά με τους αριθμούς όμως εδώ We're just checking that, that the Can we do 40 and 41 together? Although... 40 και 41 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε το 117 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 119. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μάλιστα. 119 υπέρ. Η παλιά τρόπο, η παλιά 119 έτσι. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 13α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό 13 13β υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τα δύο επόμενα καταπίπτουν 127 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ 132 να την ελέγξουμε παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 11-10 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας τώρα 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μια πρόταση να ψηφίσουμε από κοινό από το 46 έως το 3 συμφωνείτε υπέρ έως και 48 όχι όχι όλα μαζί δεν γίνεται να ψηφίσουμε αυτά 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 2 παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 13 8 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, 4, 51, 6, 5 και 6 και άλλα και το 7 και το 52 και το 8 όλα αυτά από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβασμός 2 υπέρ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 εγκρίνεται 14-7 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 67 παρακαλώ. Όχι, όχι, είναι σαφή τα πράγματα, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται την ψηφοφορία στο 67 λέει πρόεδρος ψηφοφορία, ψηφοφορίας απορρίπτεται 11-9 68 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και την 68 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία, απορρίπτεται 12 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 αποσύρθηκε. 20 Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός, ε, ε, μάλλον 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές, όχι, να ελέγξουμε το συμβασμό 8 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 13-8. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, το 87. Ψηφίζουμε από κοινού 88, 23, 24 και 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 89 παρακαλώ η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και την 90 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 12-9 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ να ελέγξουμε και την 93 άρχιτη ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 με 2 εποχές. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 υπέρ, 1 κατά. Ε, συγχαρητήρια Ελένη. So who does discharge commission? Okay, colleagues. Συνάδελφοι, περνάμε στην απαλλαγή. Νέρις, Ντέβα, κάπου τον είδα νωρίτερα. Είναι ακόμα εδώ. Α, έφυγε. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο, γιατί ο Νίρη ήταν ο εισηγητή. αν όχι ψηφίζουμε. Ξεκινούμε τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά, απόχέ. ελέγχουμε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Το προς 8 εγκρίνει. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 2, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 11 προς 7 εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 3, ψηφοφορία. Πέρας. 12 προς 8 εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Ελέγχεται 11 προς 10. Ε, συγγνώμη, εγκρίνεται 11 προς 10. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τοπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε τη 10, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ναι, ναι. 13 προς 2 και 6 αποχές. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 11 άρχεται η ψηφοφορία closed. Πέρασε. Εγκρίνεται 11 προς 10. Τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης με ηλεκτρονική ψηφοφορία ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν 16 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, τέσσερις αποχές. Ευχαριστούμε τον Έρς περνάμε στο σημείο 13. Απαλλαγή σε ό,τι αφορά το 81, το 10ο και 11ο ετά. εισηγητής είναι ίδιος, δεν είναι εδώ. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ, κατά. Ελέγχουμε την ενάρχητη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 13 προς 8, τροπολογία 2 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε την τριάρχη τριάρχητη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 12 προς 9. Τροπολογία 4 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές Έλεγχο μεγαλύτερα την 6 αν και νομίζω ότι εγκρίνεται Votes closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 12 προς 9. Τροπολογία 7 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές, ίδια διαφορά ψήφων. 8 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται το ίδιο 9 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 9 αν και νομίζω η διαφορά ψήφων είναι πέρας ψηφοφορίας 11 προς 9 πράγματι τροπολογία 12 υπέρ α, συγγνώμη τη 10 την ξέχασα υπέρ κατά αποχές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 Α, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 11 προς 9. Τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Λόγω των αποχών βέβαια νομίζω ότι εγκρίνει. Πέρασε ψηφοφορίας. Ναι. 10 υπέρ 7 κατά 4 αποχές. 20 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 18 ψήφι υπέρ. Καμία ψήφος κατά τρεις αποχές. Ευχαριστούμε τον Νέρζ. Και τώρα περνάμε στο σημείο 14, που είναι η εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΜΠ. Φρανκ Έγκελ, ε, εισηγητής, θέλετε να πείτε κάτι. Ούτως ή άλλως ε, εγώ το πήρα από ε, τον Βέντα όταν ακόμα ήταν εδώ. Νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στην διαδικασία και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. 21 υπέρ, 0 ε, κατά, δεν ξέρω κάτι. Κάποιο λάθος έγινε. Ναι, γιατί εγώ δεν είδα κανέναν να σηκώνει το χέρι του. Κάτι πρέπει να κάνετε. Να σηκώνετε τα χέρια σας καλά. 5 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 14 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η 11 υπέρ 10 κατά. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 21 άρχεται. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. 11 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 ε, με ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση επί του πρώτου τμήματος της τροπολογίας 24 άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας και εγκρίνεται 11 υπέρ 10 κατά. Δεύτερο τμήμα της 24 υπέρ κατά. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται 11 υπέρ 10 κατά. Τροπολογία 29, τροπολογία του Φρανκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την τροποποιημένη γνωμοδότηση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, μία αποχή και καμία ψήφη εναντίον. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ε, στείλουμε βέβαια και ένα σχετικό μήνυμα στην Πολωνία στον Πόγκταν. Ε, λοιπόν, σημείο 15, εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή τη δασική νομοθεσία κυβέρνηση και εμπόριο. Γιάνν ε, Ζαραντήλ, δεν τον βλέπω όμως, δεν είναι εδώ ο Γιάννη Ζαχαντήλ. Εδώ απλώς ψηφίζουμε με μία και μόνη ψηφοφορία. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την... Ε, Item 15 on the ascent. So all, so we do by Ψηφίζουμε τη συνένεση πρώτα απ' όλα. Η ηλεκτρονική ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εθελοντική συμφωνία, για την επιβολή δασικής νομοθεσίας κλπ. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Και τώρα είμαστε στο 16, είναι το ίδιο, αλλά με, την, με το ψήφισμα της συνένεσή μας. Ένα, τροπολογία 1, υπέρ, κατά. Φράγκησε υπέρ ή κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές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 Τροπολογία 17 καταπίπτει και ψηφίζουμε επομένως την τροποποιημένη γραμμοδότηση, άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασα και εγκρίνεται με 21, ομόφωνα 21 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος εναντίον. Ε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία γιατί μετατέθηκαν για το Φεβρουάριο οι επόμενες τροπολογίες, ή ε, η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ε, λοιπόν, τώρα έχουμε το ραντεβού με τη Ρουμανική Προεδρία στις 11. Δεν μπορούσαν να έρθουν πιο νωρί. Παρακαλώ λοιπόν στις 11 να είστε εδώ και μην λησμονήσετε ότι το απόγευμα έχουμε εδώ τον Επίτροπο. Να μην λείψει κανείς. Okay, colleagues. We're now moving on to item 20 on our... Συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 20 της ημέρας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον Τεοδόρ Μελεσάνου. Πες, Μελεσκάνου, μάλιστα, Μελεσκάνου, να το πούμε και σωστά. Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας. Η Ρουμανία ανέλαβε την Προεδρία στην αρχή του μήνα όπως γνωρίζουμε όλοι μια χώρα η οποία προσχώρησε το 2007 είχα μια συνάντηση με τους, τους πρόεδρους των Επιτροπών ε, πριν τα Χριστούγεννα συνάντησα και τους αδέλφους σας φαίνεται πολύ αποτελεσματική η Προεδρία σας έχουμε μια αίσθηση έτσι, δυναμισμού και ελπίζουμε βεβαίως αυτό το εξάμεινο για το Κοινοβούλιο είναι κάπως κουτσουρεμένο λόγω των εκλογών, αλλά ελπίζουμε να έχουμε έτσι μια καλή και θετική σχέση. Παραδοσιακά, συνάδελφοι, μιλάμε κυρίως για ανθρωπιστική βοήθεια εδώ σε αυτές τις συνεδριάσεις, διότι η, η εκπρόσωπος ε, είναι υπεύθυνη ε, για τα ζητήματα ανάπτυξης. Όμω εδώ έχουμε την υπόλοιπη εξωτερικών της Ρουμανίας, ο καλύπτει πολλά και διάφορα θέματα. Ήμουν το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη στην, στο φόρουμ ψηλού επίπεδου για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη και συνάντησα κάποιους, κάποια μέλη τη κυβέρνησή σα και συζητήσαμε πω ε, η Ρουμανία προσπαθεί να πετύχει του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ε, είναι πολύ καλό ότι βρίσκεστε λοιπόν εδώ σήμερα μαζί μα και περιμένουμε να ακούσουμε τι έχετε να μα πείτε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλά τα, ζητή, τα ζητήματα την Πέμπτη έχουμε μια ειδική συνάντηση για την Ιεμένη και την, κατά... και την κρίση εκεί. Συζητήσαμε και τη Βενεζουέλα, το τι συμβαίνουν εκεί, όπου καταραίει η οικονομία. Ως Επιτροπή παρακολουθούμε βέβαια και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πρόσφυγες, τις προσφυγικές ροές ανά τον κόσμο ε, και στην Ευρώπη. και έχουμε ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα σε ζητήματα ε, εκπαίδευσης για τα παιδιά ε, που βρίσκονται ε, σε στρατόπεδα προσφύγων ή που είναι σε οικογένειες προσφύγων διότι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πλέον δεν ζουν εκεί για ένα ή δύο χρόνια ζουν πολύ περισσότερα χάνουν λοιπόν την εκπαίδευσή τους όλη την εκπαίδευσή τους κάποια παιδιά προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε σε την επίκουσα κατάσταση κύριε Υπουργέ σας δίνω το λόγο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους συναδέλφους και τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι τιμή μου που μιλώ εδώ μπροστά σας σήμερα. Η Επιτροπή σας εργάζεται σκληρά και μας υπενθυμίζει τις μεγάλες ανησυχίες της εποχής μας ε, για την ευημερία της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο οι προκλήσεις είναι πολλές. Οι εκθέσεις θεωρούν ότι 132 εκατομμύρια άνθρωποι από 42 χώρες θα χρειαστούν διεθνή ανθρωπιστική αρρωγή. περισσότερε από αυτέ τι καταστάσει έχουν δημιουργηθεί από διατροφική ανασφάλεια και από ένοπλε σειράξει. Αναφερθήκατε στην Ιεμένη και στο τι θα γίνει το απόγευμα. Η Ιεμένη συμβολίζει όλη την περιπλοκότητα και την ένταση της σημερινής κρίσης, της, της κρίση ε, κρίσης, ε, ένοπλη σύραξη, ε, καταραίουν οι δημόσιες υποδομές, 20 εκατομμύρια άνθρωποι με μεγάλα προβλήματα διατροφής και βεβαίως ε, η UNICEF μας λέει και αυτό είναι σοκαριστικό σύμφωνα λοιπόν με τη UNICEF κάθε 10 λεπτά ένα παιδί πεθαίνει στην Ιεμένη είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα των ε, τεράστιων διαστάσεων ε, των παίρνει μια ανθρωπιστική κρίση σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως η ένοπλη στην Συρία έκτη χρονιά πολέμου χωρίς να φαίνεται να υπάρχει μια προοπτική για μια επιστροφή των κατοίκων εκεί κοντά στην Ασία, στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ευρώπη πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την ένοπλη σύραξη εκεί. Έχει οδηγήσει αυτό σε μετατόπιση πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων. Και 3,4 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι εκεί χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Οι φυσικέ καταστροφέ, όπω στην περίπτωση, τη Ινδονησία, επίση έχουν οδηγήσει ε, σε μεγάλη ζημία Συγγνώμη για αυτή την εισαγωγή, την κάπως απότομη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να την αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, αναμένεται, να είναι, αναμένεται από αυτήν να είναι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ενίσχυση και την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Όπως τα γνωρίζετε, η Ρουμανία θεωρεί ότι η συνοχή αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματός μας. Η εσωτερική συνοχή αλλά και η εξωτερική συνοχή. Και αυτό με οδηγεί στην δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Είναι η ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος παίκτης. Με όλες ε, τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή. Είναι υποχρεωμένη να αναλάβει τις ευθύνες της. Η ανθρωπιστική βοήθεια, οι πολιτικές συνεργασίες για την ανάπτυξη είναι εργαλεία για να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος παίκτη, αφήνοντας πίσω την ιδέα Όχι, κάποιο τηλέφωνο πρέπει να ήταν. Δεν έχει σχέση με την Επιτροπή μας πάντω. Μήπως είπα κάτι που δεν έπρεπε να πω, λέει ο υπουργό. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στις προτεραιότητες της Προεδρίας μας και το πρόγραμμά μας και να μιλήσω και για συγκεκριμένες δράσεις είναι προφανές ότι ο δρόμος που οδηγεί στη λύση συχνά ξεκινάει από την πρόληψη. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η Ρουμανία θα δώσει έμφαση ως πρώτη προτεραιότητα τον ρόλο της μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Διαχείριση, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Η Προεδρία μας θα επικεντρωθεί λοιπόν και στη διαδικασία εφαρμογής. Επιπλέον θέλουμε να δημιουργήσουμε δυνατότητες για άμεση ιατρική απάντηση. Είναι πολύ βασικό αυτό για να μπορέσουμε να λύσουμε, να συσσώσουμε ζωές όταν διαχειριζόμαστε κρίσεις. Ταυτόχρονα θα εθαρρύνουμε την διασύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής ενίσχυσης και των, ε, της πολιτικής προστασίας και των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα με το πλαίσιο ασφάλειας ε, και τα συμπράσματα του Συμβουλίου για την εκπαίδευση κατά της κρίσεις και τις επίγουσες καταστάσεις θα δοθεί έμφαση στον ρόλο της εκπαίδευσης, στην προώθηση της μείωσης του ρίσκου και την αθεκτικότητα. Η εκπαίδευση στα κέντρα προσφύγων, όπως είπατε, ε, είναι το κλειδί για τον μέλλον μας, ε, διότι εκεί δίνουμε έμφαση στα παιδιά, στους νέους. Αυτοί εκπροσωπούν μιας πιο ευάλωτες ομάδες όταν προκύπτει μια κρίση, καθώς μεγαλώνουν σε ένα πλαίσιο που συχνά ε, επηρεάζει αρνητικά την εκπαίδευσή τους, τη μόρφωσή τους. Πρέπει να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο να χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Να τον αποτρέψουμε. Η έγκαιρη προειδοποίηση, η προετοιμασία βοηθάει στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εκπαίδευση σε περίπτωση κρίση και καταστροφή. Χρειαζόμαστε ισχυρά συστήματα συμπράξει για μια γρήγορη, αποτελεσματική και καινοτόμο απάντηση σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω τι ιδιαίτερε ανάγκε των αγοριών, των κοριτσιών, των ανθρώπων με αναπηρία. Μια πολύ σημαντική πτυχή που δημιουργεί σημαντικέ συζητήσει είναι η οικονομική πτυχή η δυσκολία χρηματοδότησης ε, στον τομέα αυτών έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις με κάθε δωρητή, μεταξύ υπάρχει μακροπρόθεσμη πρόληψη, υπάρχει η άμεση ανταπόκριση. Ε, στην εντολή μας θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους, στην θητεία μας, να βρούμε τρόπους έτσι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τα σχετικά κονδύλια να μπορέσουν να πάνε προς πρωτοβουλίες στον τομέα αυτών. Έχει την ε, ε, το καθήκον Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια προβλέψιμη απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Πρόσφατα εορτάσαμε το νέο έτος, ε, κυρίε και κύριοι, μια χρονιά που ανήκει σε μια εποχή όπου τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Αυτό μας δίνει πολλές ευκαιρίες, ταυτόχρονα όμως έχουμε μπροστά μας και πολλές προκλήσεις. Και μία από αυτές έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες. θέλω να πω δύο λόγια για τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες θεμελιωδώς αλλάζουν τον κόσμο, τον κόσμο μας και ο ανθρωπιστικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση. Εδώ μιλάμε για drones, για τεχνητή νοημοσύνη, για εφαρμογές τεχνητής ε, πραγματικότητας, εικονικής πραγματικότητας. Όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν ή ε, να ε, δυσχεράνουν την αρρωγή και τη συνδρομή. Συζητούμε λοιπόν με τι διάφορε βλεγόμενε φορεί, έτσι ώστε εμεί, ω δωρητέ, να βρούμε τρόπου να συνεισφέρουμε η καινοτομία αυτή ε, να βοηθήσει ε, στον ανθρωπιστικό τομέα. Είτε μιλάμε, τομέα, είτε μιλάμε για φυσικέ καταστροφέ, είτε μιλάμε για ενόπλε σειράξει. Ο στόχο είναι διτό. Πρώτον, πώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι τεχνολογίε για να μπορέσει να φτάσει η βοήθεια καλύτερα σε αυτούς που πρέπει να φτάσει και πώς οι δικαιούχοι θα μπορέσουν στη συνέχεια να απορροφήσουν καλύτερα αυτή την βοήθεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες ε, στον τομέα της ανθρωπιστικής καινοτομία με τον ιδιωτικό τομέα προωθώντας ένα δίκτυο ε, με σημεία εστίασης ε, όπου συμμετέχουν κράτη-μέλη, διοικήσεις, ο ιδιωτικός τομέας. Είναι κάτι το οποίο έχει προσχεδιάσει η Κομισιόν από κοινού με τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καινοτομία από μόνη της δεν είναι πανάκια. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προσεκτικά. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με τις νέες αυτές τεχνολογίες όπως αυτοί που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τη διάδοση ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τι επιπτώσει για του πολίτε και του ανθρώπου που εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα όταν νέε τεχνολογίε όπω ε, τα drones χρησιμοποιούνται σε, πολεμ, σε πολεμικές σειράξεις ή ε, σε ε, αποστολέ αναζήτηση και διάσωση. Υπάρχει ομάδα εργασία για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διατροφή. πρέπει να γίνει μια δουλειά λοιπόν στο ότι θα ιδιαίτερα την παρακολούθηση ανθρωπιστικών κρίσεων Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν στενά μια σειρά από ανθρωπιστικέ κρίσει που είναι εξελίξει, που, είναι, που θα είναι μελλοντικέ ή που κρατούν εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο από κοινού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες πόρους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Προεδρία θα προωθήσει με τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, την Κομισιόν, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και βεβαίως ε, θα είμαστε και στενά ε, συνδεδεμένοι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα καλέσουμε τρίτους, όπως εκπροσώπους ε, από τη Διεθνή Κοινωνία των Πολιτών και τις σχετικές οργανώσεις για να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους, την εμπειρία τους. Δεδομένου του εύρους της παρούσας κρίσης και επειδή αυτή, οι αιτίες της κρίσης είναι μικτές, μία ένοπλη σύραξη μπορεί να συνδέεται με την ξηρασία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διατροφική κρίση, κρίση μέσα στην κρίση δηλαδή. Ε, και υπάρχει επίσης ε, όλο και μεγαλύτερη ε, παραβίαση των, της ανθρωπιστικής νομοθεσίας. Είναι λοιπόν πολλή δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Κάτι ακόμα, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι σειράξεις. προχωρούν. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια πιο συνεπή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, ανθρωπιστική ε, βοήθεια και την ειρήνη. Δεν μπορούμε ε, να το πετύχουμε αυτό αν δεν έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, πιο σφαιρική ευρωπαϊκή προσέγγιση όπου ενώνουμε τι δυνάμει μα και πολλαπλασιάζουμε τον αντίκτυπο των προσπαθειών μα. Η Ρουμανική Προεδρία δεσμεύεται να δώσει έμφαση έτσι ώστε να εφαρμοστεί αυτό από κοινού με την πολιτική συμφωνία του 2017 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως αυτό αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Συνένεση, στο Ευρωπαϊκό Κονσένσου για την Ανάπτυξη. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να Έχουμε μια επιτυχή διαπραγμάτευση της εταιρική σχέσης μετά το Κοτονού. Εμείς συχνά λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Συνεργασία με μια μεγάλη ομάδα χωρών ΑΚΕ ως συνεισφορά της Προεδρίας μας σκοπεύουμε να οργανώσουμε την 37η Σύνοδο ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή κοινοβουλευτική σύνοδο στα τέλη Μαρτίου στη Ρουμανία. Ελπίζουμε αυτό να οδηγήσει σε χρήσιμες συζητήσεις για την ενίσχυση ε, της τωρινής αλλά και της μελλοντικής αυτή εταιρικής σχέσης. Κυρίε και κύριοι, θεωρώ ότι είναι σημαντική η συνάντησή μας. Ε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος που να ξεκινήσει μια προεδρία από το να ξεκινήσει ένα διάλογο με τους ε, εκλεγμένους εκπρόσωπους του ευρωπαϊκού λαού. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική διαθεσμική συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Είμαι λοιπόν διατεθειμένο και προσωπικά να συνεργαστώ με την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, με τον καθένα από εσά. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με ακούσατε, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω εδώ και περιμένω τα ερωτήματά σας και έναν ζωντανό διάλογο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την επισκόπηση αυτή μας παρουσιάσατε και με χαρά άκουσα να λέτε ότι οι Υπουργοί ενδιαφέρονται για την ε, παρατεταμένη αυτή κρίση που πάνω από πέντε χρόνια τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες χώρες. Ε, η ανθρωπιστική βοήθεια φυσικά και δεν πρέπει να λάβει πολιτικό χαρακτήρα. Χρειάζονται πολιτικές λύσεις βέβαια στις κρίσεις αυτές, γιατί τόση εξαθλίωση δεν μπορούμε να τη δεχθούμε. Στον κόσμο σίγουρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα και της κλιματικής αλλαγής, αλλά η εξαθλίωση σε πολύ μεγάλο βαθμό προκαλείται από την ανθρωπότητα την ίδια και χρειάζονται πολιτικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σταθερά βοήθεια. Είχαμε με το δίκτυο ΜΚΟ Voice ε, μια συνάντηση ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας και μας ζήτησαν να, να βάλουμε περισσότερη ενέργεια για την πολιτική αντιμετώπιση των παρατεταμένων κρίσεων, γιατί πρέπει να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις, αλλιώς δεν θα ε, πάψουν να υπάρχουν αυτές οι Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση ο κύριος ε, Φρουντζούλικα καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη χαρά μου που καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μελεσκάνου. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησα ε, το, τη δεκαετία του 90 τη σταδιοδρομία μου όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Μελεσκάνου. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Ήταν λοιπόν τότε Υπουργό Εξωτερικών, έχει διατελέσει τρει φορέ Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Εθνική Άμυνα, έχει διατελέσει και άλλα ε, πολύ σημαντικά αξιώματα. Είχε. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν κύριε Υπουργέ, είστε ένα εξέχων διπλωμάτη, χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Μετά την παρέμβασή σα θα ήθελα ένα σύντομο ερώτημα μόνο να σα υποβάλω. Για παράδειγμα, πώς βλέπετε τη Ρουμανική Προεδρία ε, και την ε, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει. Σίγουρα γνωρίζουμε την ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτά τα δύο ε, πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το εξάμεινο της Προεδρίας σας και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ σήμερα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω και σας συγχαίρω που ε, έχετε εκλεγεί ευρωβουλευτή. Ελπίζω μετά τις εκλογές στα τέλη Μαΐου να επανέλθετε και να συνεχίσετε, συνεχίσετε να είστε ένας από τους πολύ δραστήριους ευρωβουλευτές εδώ. Θα να σας ευχαριστήσω για το ερώτημά σας πολύ φιλικά μου το θέσατε, αλλά είναι πολύ δύσκολο παρόλα αυτά το ερώτημα, διότι στην πράξη η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες ε, για την αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημάτων. Κατά την άποψή μου, ποιος είναι ο μόνος λογικός τρόπος να προχωρήσουμε πρέπει να συνδέσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια αφενός με την αναπτυξιακή βοήθεια αφετέρου. Αν θέλουμε πραγματικά να συμβάλλουμε ε, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χρειαζόμαστε κονδύλια, χρειαζόμαστε έργα, project, ώστε οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που είναι αντιμέτωπες με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής να μπορέσουν την οικονομία τους, να την απομακρύνουν από το σύστημα κατανάλωση άνθρακα στις ε, ενέργειες τις πιο καθαρές, αιωλική, ηλιακή κτλ. Και η δική μας Προεδρία πρέπει να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δηλαδή η πολιτική μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ απλή. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας πολύ ζωντανός, ανοιχτός διάλογος. Να δοθούν σαφείς δεσμεύσεις ε, και να γίνει λόγος για συγκεκριμένα έργα, project. Το ίδιο ισχύει και για τη μετανάστευση. Όλοι ανησυχούμε και αναζητούμε τρόπους να σταματήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα. Και από την αρχή η Ρουμανία είχε επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια, η ρίζα του προβλήματος, που είναι δύο τεινά. Τα προβλήματα αυτά είναι η εσωτερική, η πόλεμη, η εμπόλεμη σειράξη στην περιοχή και η κλιματική αλλαγή. Έξω και για εμά, η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των χωρών αυτών, αλλά και την ασφάλεια τη Ευρώπη. Γι' αυτό και είμαστε έντονα ε, υπέρμαχοι της ιδέας να υποστηριχθούν ε, έργα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος, έστω στον τομέα ε, αυτό της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν κακές ειδήσει, δεν θέλω να σας χαλάσω τη μέρα βέβαια. Ακούσαμε, νομίζω, πότε δεν ξέρω πού, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ότι αναμένεται φαινόμενο Ελνίνιο για φέτος. Αυτό είναι πολύ κακό νέο. Σκεφτείτε τα νησιωτικά κράτη, στον Ειρηνικό ή σε άλλες περιοχές. Τι θα συμβεί εκεί με τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ιδέα πως πρέπει τις χώρες αυτές να τις παροτρύνουμε, να τις στηρίξουμε για να χρησιμοποιούν πράσινες μορφές ενέργειας και ταυτόχρονα σε διεθνές επίπεδο πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις, οι παγκόσμιες δεσμεύσεις για το κλίμα. Και αυτά είναι ένα από τα λίγα ζητήματα που ούτε σε εθνικό ούτε σε περιφερειακό καν επίπεδο δεν μπορείς να βρεις λύσει Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο που αφορά όλη την ανθρωπότητα. Η δική μου γνώμη είναι η εξή Μια από τις προτεραιότητες μας ως Προεδρίας είναι να διαδραματίσουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, για την πρόθεση του πολυμερούς συστήματος, της πολυμερούς προσέγγισης. Και αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ άλλων ε, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ένωσης ε, στις ε, δραστηριότητες για το θεματολόγιο του 2030 πρέπει να είναι πολύ πιο δραστήρια σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση των διεθνών προσπαθειών. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον μόνιμο εισηγητή μας για ε, τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας στον Ενρίκε Γκερέρο Σαλό, που είναι υπεύθυνο για αυτά τα θέματα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Εμείς που έχουμε κάποια σχετική εμπειρία από συνεδριάσεις όπου έρχονται υπεύθυνοι ε, χωρών που για πρώτη φορά αναλαμβάνουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν λέω γνωρίζουμε ε, τον ενθουσιασμό και, τις, ε, και την προσπάθεια που καταβάλουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι τα καλύτερα και οπωσδήποτε ε, να υπολογίζεται και επί της βοηθείας του Κοινοβουλίου. Ε, και ε, βέβαια μετά από τον Απρίλη εμείς θα εξαφανιστούμε από την πολιτική σκηνή γιατί θα έχουμε προεκλογική εκστρατεία. Μερικοί από, από εμά, ο κύριος Φρανσουλίτσα παραδείγματο χάρη, γιατί εγώ δεν θα είμαι υπεύθυνο. Κοιτάξτε, ακόμα έχουμε βέβαια και θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον, Brexit, όχι Brexit, τι θα κάνει η Κομισιόν ε, την, ε, στην επόμενη θητεία κτλ. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένες ε, ειδικέ ε, σειράξεις Ουκρανία, Συρία, Ιεμένη, ε, κάποιες φυσικές καταστροφές όπως την Ινδονησία. Αλλά αυτό που θεώρησα πολύ ενδιαφέρον και στο έγγραφο των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας και σε αυτά που είπατε πριν από λίγο, είναι ακριβώς ε, η γενικότερη εστίαση, δηλαδή οι ε, κεντρικές προτεραιότητες ε, και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων αναφέρεται και η προσπάθεια μείωσης κινδύνου από φυσικές καταστροφές αλλά και άλλου είδους καταστροφές. Και επίσης η εφαρμογή των συμφωνιών Σεντάι και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πλατφόρμα του Κανκούν. Και για τα όσα θα συζητηθούν στις 17 Μαΐου στην ε, Γενέβη. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ, έχετε ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση για τις ε, προτεραιότητες που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και που θα υποβάλει στην συνεδρίαση της Κεντρικής Πλατφόρμας στη Γενέβη. στην πρόληψη κινδύνων και καταστροφών υπογραμμίζεται ε, την ε, ε, ανάγκη να δημιουργηθούν υποδομές υγείας στις χώρες αυτές οι οποίες περισσότερο εκτεθειμένες είναι σε κινδύνους λόγω των γεωλογικών και λοιπόν γεωγραφικών ας πούμε ειδικών συνθήκων που επικρατούν. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει εκφράσει τον προβληματισμό του ε, για τις ελλείψεις ε, υποδομών υγείας σε χώρες όπως Νότιο Σουδάν, Κονγκό, ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Προεδρία θα προσπαθήσει να εντατικοποιήσει αυτήν την στήριξη σε αυτές τις χώρες εντός του Συμβουλίου. Γνωρίζετε βεβαίως ότι το κοινοβούλιο μας ήταν ιδιαίτερα δραστήριο στην παροχή κονδυλίων για την εκπαίδευση των παιδιών ε, εν μέσω ε, κρίσεων ανθρωπιστικών και λοιπόν. Ε, βεβαίως εμείς προσδοκούμε ως κοινοβούλιο σε κάτι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μακάρι από το 6% που τώρα αφιερώνουμε στην ε, εκπαίδευση σε καταστάσεις ε, ε, κρίσεως να περάσουμε σε σε ένα ποσοστό υψηλότερο. Αυτό είναι σημαντικό για τη διασύνδεση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην ανταπόκριση σε περιπτώσεις κρίσεως και την την αναπτυξιακή βοήθεια γιατί πολλές φορές ε, κάποιες καταστάσεις κρίσεων εγκαθίστανται στις χώρες και γίνονται κρίσεις μεγάλης διάρκειας και επομένως ε, σε αυτά τα πλαίσια η εκπαίδευση αποτελεί στρατηγικό κεντρικό στόχο. Επίσης αναφερθήκατε και σε κάποια άλλα σημεία. Αναφερθήκατε στον ανθρωπιστικό νόμο, στις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και πιστεύω ότι κάθε φορά κινδυνεύει ε, όλο και περισσότερο ε, η ζωή των ε, ανθρωπιστικών, των εκπροσώπων ανθρωπιστικών οργανώσεων που δουλεύουν επί τόπου, όλο και περισσότερη γίνεται η βία απέναντι σε ανθρωπιστικές προσπάθειες και αποστολές και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να σκύψουμε πάνω στο θέμα αυτό. Τελευταίο, γιατί βλέπω εδώ και την ε, Ελένη Θεοχάρους που προφανώς θα πάρει και αυτή το λόγο γιατί ήταν και η συγγήτρια. Ψηφίσαμε σήμερα και εγκρίναμε την ε, έκθεση της ε, που αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Και στην Επιτροπή μας εκφράσαμε την άποψη ότι ένα σημαντικό τμήμα αυτού του ε, σώματος αλληλεγγύης θα πρέπει να αφορά την υποστήριξη σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής ε, κρίσης. Τέλος, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την ενημέρωση που μας κάνατε, τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και ευελπιστώ ότι ε, θα ε, τα πούμε σύντομα στην συνεδρίαση και στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ε, θα γίνει στην χώρα σας τον Μάρτιο η συνάντηση της Ισομερούς εκπροσώπηση ΑΚΕ. Ξέρουμε ότι η κατάσταση στο Κονγκό δημιουργεί προβλήματα, αλλά και στην Αγγόλα επίσης ε, είχαμε ε, ε, στην αρχή της θητείας μας την κρίση έμπολα και τι μας δίδαξε ε, αυτό είναι ότι εάν θέλουμε να μπορέσουμε ε, ε, να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως αυτή του ιού έμπολα θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να απομονώσουμε τις περιπτώσεις. Και αυτό που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι και στην Δυτική Αφρική έχουμε δώσει πολλά χρήματα, έχουμε επενδύσει πόρους ε, και δίνουμε χρήματα στη διάρκεια της κρίσης, αλλά μόλις τελειώσει η κρίση σταματάει η βοήθεια και έχεις δίκιο όταν λες ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή βοήθεια έτσι ώστε τα διδάγματα να είναι ε, διαρκή. Να απαντήσετε αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Γκυρέρο για τα ερωτήματα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι το να επενδύσει κανείς στη μείωση του κινδύνου, του ρίσκου από καταστροφές ουσιαστικά οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων και πρέπει να είναι μια σημαντική κατεύθυνση αυτή της πολιτικής μας. Αναμένουμε βεβαίως την έκτη παγκόσμια πλατφόρμα για τη μείωση των, του ρίσκου από καταστροφέ στη Γενέβη το Μάιο και έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε για την προπαρασκευή της της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάντηση αυτή της Γενέβης θέλουμε να υπάρξει μια πλατφόρμα ε, από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Εμείς θα υποστηρίξουμε οπωσδήποτε τις ε, δραστηριότητες προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα για την εκπαίδευση. Ε, πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Σε κάποιες χώρες έχουν γίνει κάποια βήματα. Συνάντησαν, ε, επισκέφθηκαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα προσφύγων ε, από τη Συρία στην, στην Ιορδανία και υπάρχουν και σχολεία εκεί ε, στο, στα στρατόπεδα, δηλαδή, αλλά αλλού, αλλού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ένα σημαντικό στοιχείο και αναφέρεται αυτό στα συμπεράσματα για την εκπαίδευση ε, για τις καταστάσεις, τις καταστάσεις κρίσης τον Νοέμβριο και εκεί υπογραμμίζεται ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Εμείς παρακολουθούμε την εφαρμογή των συμπερασμάτων αυτών. Η εκπαίδευση, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια ε, και την αξιοπρεπή διαβίωση η εκπαίδευση είναι πολύ καλή επίσης ε, για να μην ε, ζωσπαστικοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου η θρησκεία είναι διαφορετική. Ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Θα βοηθήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν, να συντονίσουν όπως πρέπει την 7η ε, διάσκεψη σχολείων που θα γίνει ε, στο Μάιο στην Ισπανία και θα προωθήσουμε και τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση νομίζω στο θέμα ε, της όντας μεταξύ των δύο φύλων, στην βία που βασίζεται στο φύλλο. Εμείς θα εξασφαλίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε στενά τα συμπέρασματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου. Αναφερθήκατε επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς θα υποστηρίξουμε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας. Είναι βασική προτεραιότητα και για μας. Σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, η απόφασή σας, ο στόχος σας, ε, να προσφέρετε 10% του για την παιδεία είναι κάτι που θα το υποστηρίξουμε ως πρόταση από κοινού αδέλφους ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και συζητήσεις για να επιτευχθεί πλειοψηφία προς αυτήν την κατεύθυνση. Λάβαντα υπόψη βεβαίως και τις θέσεις άλλων κρατομελών θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε όπως είπα και με το κοινοβούλιο στο σύνολό, της, στο σύνολό του διότι είστε κινητήριος, ο κινητήριος μοχλός για την πρόθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Είναι... Ευχαριστώ και αυτό που είπατε για τον προπολογισμό είναι ευπρόσδεκτο. Ο Πίτροπο Τηλιανίδη θα έρθει και σήμερα το μεσημέρι και έχει εκδώσει ένα, μια ανακοίνωση τύπου ε, που μιλά για 1,6 δι που είναι το ψηλότερο ποσό για ανθρωπιστική βοήθεια. Αρχικώ. Ε, είναι η λέξη σημαντική. Γιατί πολλές φορές ε, δεν διαθέτουμε το επαρκές ποσό και αρχίζουμε να προσθέτουμε στη διάρκεια του έτους. Ε, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι κάνουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να χειριστούν τα κονδύλια. Είτε κάποιος από τη Βόρεια Ουγγάντα και αυτοί παίρνουν πρόσφυγες από το, από Νότιο Σουδάν και τον Ιανουάριο τους δίνουν χίποσο. Και έπειτα τους δίνουν λίγο παραπάνω και πρέπει να ζητούν συνεχώ νέα χρηματοδότηση. Άρα το επιτόπιο προσωπικό ουσιαστικά ζητά χρήματα. Εκεί ε, χάνει πολύ χρόνο και προσπάθει για να συμπληρώνει αιτήσει, για να ζητά συμπληρωματική χρηματοδότηση. Και δεν μπορούν να προγραμματίσουν. Ξέρουμε τι γίνεται ε, στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν και πότε θα λυθεί και το πρόβλημα. Ελπίζω το Συμβούλιο να κατανοήσει το πρόβλημα. Εμεί ε, έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει τη σημασία που έχει να δοθεί αρχικά ο επαρκή προπολογισμό για να μπορούν επιτόπου ε, να κάνουν τον προγραμματισμό Έχουμε και το πολιετές, τις πολιετέ δαπάνες, δεν πρέπει να το χάσουμε. Θα ρωτήσουμε και τον Επίτροπο Ενρίκη. Γίνεται λόγος για ένα τριετή προγραμματισμό και όχι η ετήσια χρηματοδότηση. Ακούσαμε σε μια άλλη συζήτηση, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω στο Μαλί, η ανθρωπιστική βοήθεια γιατί εστιάσαμε ξαφνικά ή στον Ήγηρα. Τέλο πάντων, υπήρχαν περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση, ε, για ανθρωπιστική βοήθεια και ε, απ' την άλλη είχαμε τη μακροπρόθεσμη πολιτική και αυτά δεν ε, ταιριάζουν κατά κάποιο τρόπο. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θα δούμε τι θα γίνει στη νέα περίοδο. Ελπίζουμε με τα προγράμματα να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ελλήνη Θεοχάρου γιατί ακούσαμε δύο σοσιαλιστέ. Έχετε και εμπειρία από ανθρωπιστική βοήθεια, θα μας τα πείτε καλύτερα. Κυρία Πρόεδρε, Mr. Minister, I will speak. Θα μιλήσω ελληνικά, ε, κύριε Πρωθυπουργέ. Thank you. Ε, θα ξεκινήσω από εκεί που ε, τελείωσε ο κύριος Γκερέρο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, νομίζω ότι το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός στόχος αυτού του σώματος είναι να αναπτύξει ανάμεσα στους νέους της Ευρώπης το αίσθημα και την ευθύνη και την υποχρέωση της αλληλεγγύης απέναντι σε αυτούς που είναι λιγότερο τυχεροί, απέναντι σε αυτούς που δεν θέλουμε να τους αφήσουμε πίσω. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Υπουργέ για το όραμα το οποίο μας έχετε παρουσιάσει. Είναι πράγματι ε, μεγαλειώδες αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και την ε, προσπάθεια που θα καταβάλει η Ρουμανική Προεδρία προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Ρουμανία αντιμετωπίζει ίδια οικονομικά προβλήματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παίρνει πρωτοβουλίες κάποιος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει ακριβώς η ανθρωπιστική κρίση. Θέλω να διαχωρίσω ξεκάθαρα την ανθρωπιστική κρίση και τη βοήθεια που παρέχουμε εκείνη τη στιγμή που υπάρχει ανθρωπιστική κρίση από την ανθρωπιστική βοήθεια που είναι άμεσα συνειφασμένη με την αναπτυξιακή βοήθεια. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια μπορούν να συσχετιστούν. Αλλά η κρίσιμη στιγμή όπου άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, για παράδειγμα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν μπορεί να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω ποιοι έχουν κάποιες ανάλογες εμπειρίες, τι ε, λογής ε, ανάπτυξη θα σκεφτείς όταν για ένα παιδί δεν έχεις ε, δύο δράμια νερό να του δώσεις για να μην πεθάνει από την αφυδάτωση. Γι' αυτό το λόγο και γνωρίζοντας ότι μέσα στην Ήπειρο μας, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλοί πληθυσμοί που ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας ε, και στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη όπου υπάρχουν συσσωρευμένοι πρόσφυγες, φυγάδες που έχουν φτάσει στην Ευρώπη. Μην νομίζετε ότι με το που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως έχουν λυθεί τα προβλήματα τους. Περνούν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά και οι χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση έχουν πληθυσμούς που ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας και καταβάλουμε υπέρμετρες προσπάθειες για να τους κρατήσουμε σε μια ε, ε, περιοχή όπου γυτνιάζει θα μπορούσε να πει κανείς με την επιβίωση. Το ίδιο συμβαίνει και για μετακινούμενους πληθυσμούς μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία χώρα στην άλλη ελπίζοντας σε μια καλύτερη ζωή. Στον άμεσο περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι μαστίζονται από φοβερά προβλήματα, από την πείνα, την υποανάπτυξη, την έλλειψη υποδομών, την εγκατάλειψη κυρίως από αυτό το ότι τους έχουμε ξεχάσει. Είναι οι Παλαιστίνοι οι πρόσφυγες που ζουν στους Παλαιστινιακούς οικισμούς του Νοτιού Λιβάνου. Είναι η Γάζα. Είναι η Εμένη που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να αναπτυχθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος και να μην πεθαίνει κάθε 10 λεπτά ένα παιδί στην Εμένη. Να πηγαίνουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα τα οποία κατά τα άλλα εφόσον δεν έχουμε ευρωπαϊκά να ρίχνουν τρόφιμα μέσα στην ε, χώρα αυτή είναι το ότι συμβαίνει στη Συρία και στις περιοχές της, ε, του Κουρδιστάν οι οποίες υφίστανται την πολεμικέ τις πολεμικές επιπτώσεις πολλών που έχουν σπέσει εκεί πέρα τα χαμδίθεν για να φέρουν την ειρήνη αλλά στην πραγματικότητα για να ελέγξουν τις οδούς του πετρελαίου. Είναι τα 12 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι συνοστισμένοι στην Λιβύη και προσπαθούν να φτάσουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στα χέρια διαφόρων συγχρόνων ε, δουλεμπόρων και είτε πεθαίνουν από την πείνα είτε πνίγονται μέσα στις ε, θάλασσες. Για αυτούς τους λόγους, αν η Ρουμανική Προεδρία αναλάβει μια πρωτοβουλία να λυθεί αυτό το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, να σώσουμε όσο το δυνατό περισσότερες ζωές, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε παραπέρα και για ανθρωπιστική βοήθεια και για αναπτυξιακή βοήθεια. Και πάλι σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Υπουργέ και θέλω να εκφράσω τον ε, μεγάλο θαυμασμό μου για την ε, χώρα σας και τον λαό σας. Ευχαριστώ. Thank you. Well, um, you gave us a big, many countries, Minister. Merci. I don't know if you have some responses. Δεν ξέρω αν έχετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις, ε, κύριε Υπουργέ. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Θεοχάρους. Πρέπει να σας πω πολύ ειλικρινά, κύριε Θεοχάρους, ότι αγγίξατε κάποια από τα πλέον ε, λεπτά και εύθραστα σημεία της ε, πολιτικής και των δραστηριοτήτων μας. Αναφερθήκατε σε διάφορες ε, περιπτώσεις, μετανάστες, πρόσφυγες, ε, χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ δυσχερή κατάσταση λόγω πολέμου, η Εμένη, η Συρία και άλλα. Θα ήθελα να σας πω ότι μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ρουμανίας ήταν η δημιουργία το 2017 μιας επίσημης οργάνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας, ενός φορέα λοιπόν που προωθεί και χρηματοδοτεί έργα, αναγνωρίζω ότι εστιάζει κυρίως στο, στη Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, στα Δυτικά Βαλκάνια. Εντάξει, δεν είναι και τέλεια, αλλά είναι ε, μια εξειδικευμένη οργάνωση η οποία συνδυάζει την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή βοήθεια. Φέτος, μάλλον όχι, πέρυσι, έγινε ε, δεκτή σε επίπεδο ΣΑ, σε μια ειδική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορες χώρες στο Παρίσι. Δεν συζητούμε λοιπόν μόνο, αλλά εγκρίνουμε στην πράξη μέτρα και ενθαρρύνουμε τους διάφορους ε, φορείς να συμμετέχουν στις σχετικές προσπάθειες ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Ναι, υποδεχόμαστε πρόσφυγες και πριν δύο εβδομάδες μάλιστα από την Ιταλία. Όχι, από τη Μάλτα, από τη Μάλτα. Όμως και εμείς αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση με εσάς, υπό την έννοια ότι αυτοί που θέλουν να είναι πρόσφυγες δεν ενδιαφέρονται και τόσο να παραμείνουν στη Ρουμανία, αλλά τη θεωρούν ως χώρα διέλευσης, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να φτάσουν τελικά σε μια χώρα όπου κοινωνικέ υπηρεσίε, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, είναι πιο γενναιόδρε, οι βόρειε σκανδιναβικέ χώρε, στη Γερμανία ή αλλού. Εκεί θέλουν να φτάσουν. Εμείς συνεχίζουμε όμως να τους υποστηρίζουμε και να τους προσφέρουμε την προοπτική, αν θέλουν να κατασταθούν. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σωμαλή Λεγγύης, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και ειλικρινά Θέλω να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερω τι προσπάθειες τη Αυστριακή Προεδρίας που δρομολόγησε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε, να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε να προχωρήσουμε αυτό το φάκελο λοιπόν και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν οι τριμερείς οι οργανικές διαβουλεύσεις και να εγκριθεί στο δικό μας εξάμεινο. Τώρα, κατά τα λοιπά. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο στη διάθεσή σα, σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Το πρωί ψηφίσαμε την έκθεση τη κυρία ε, Θεοχάρου ακριβώ για το ε, σώμα αυτό αλληλεγγύη και μακάρι να περάσει ε, και να έχουμε τον τριμερή διάλογο. Νόρμπερτ Νόιζερ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και τον κύριο Τσέλερ που έχει ζητήσει το λόγο. Ο Νόρμπερτ καταρχάς όμως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στην ε, συνεδρία της Επιτροπής μας. Είστε πολύ ε, πεπειραμένος στην πολυμάτια, όπως είπε και ο Ντούρου Για μας το κοινοβούλιο είναι λίγο πιο εύκολο να μιλάμε ξεκάθαρα. Ήθελα λοιπόν να κάνω μια δήλωση για το τι έκανε η Κομισιόν πριν αναλάβετε την Προεδρία. Δεν ήταν δίκαια τα σχόλια, διότι στην αρχή, αλλά και πριν ακόμα, είχατε δείξει ότι διέπεστε από πολύ ευρωπαϊκό πνεύμα. Και θα το καταδείξω αυτό με κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Το Δεκέμβριο είχαμε τη συνάντηση Κοτονού, ε, ακέ στο Κοτονού. Υποτίθεται ότι η Αυστριακή Προεδρία έπρεπε να δραστηριοποιείται. Αλλά αρνήθηκαν με κάποιο τρόπο, οπότε αναλάβατε εσείς. Και ήταν εκεί η σας, ε, μια γυναίκα συγκεκριμένα, πολύ εντυπωσιακά αυτά που έλεγε και πραγματικά η προσπάθεια και η προσήλωσή της για τα θέματα ΑΚΕ και στην Προεδρία σας όπως αναφέρατε θα βοηθήσετε η εταιρική σχέση κοτονού να περάσει στο επόμενο στάδιο. Αυτό ήταν πολύ θετικό που το υπογραμμίσατε. Και θα θέλαμε να συνεργαστείτε και με την Προεδρία που θα σας ακολουθήσει, τη Φινλανδική. Και εμείς βέβαια θέλουμε να συνεισφέρουμε. Επίσης το Μάρτιο θα φιλοξενηθεί η ε, συνέλευση τη εκπροσώπησης και Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ζινάγια στην Ρουμανία. Κάποια κράτη-μέλη κατά το παρελθόν, ξέρετε, είχαν αρνηθεί κιόλα να συνεργαστούν στενότερα με τους εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ. Άρα σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να τονίσω είναι ότι νομίζω είστε η μόνη νοτιευρωπαϊκή χώρα που υποδέχεται πρόσφυγες από τη Μάλτα λόγω της κρίσης που έχει προκύψει. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να διαπιστείτε από το ευρωπαϊκό αυτό πνεύμα και να γνωρίζετε επίσης ότι εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, και η αναπτυξιακή πολιτική σε σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο. Μιλήσατε για την ανθρωπιστική βοήθεια επίσης και για την αναπτυξιακή πολιτική πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Νομίζω ότι η ίδια πολιτική φιλοσοφία μας εμπνέει και εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη δέσμευση που δείχνετε για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. now it's working. Yeah, now it's working. Thank you very much, Mr. Neusser. It's, it's a pleasure to have such a question because it's one of the priorities of, of, of our presidency. We assumed from the very beginning the idea that... Είναι μια σωτερότητα της Προεδρίας μας και ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Μιλάμε τώρα για χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού, τη Συμφωνία του Κοτονού, ε, που χρειάζονται αυτή την βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Εμείς ε, αναλαμβάνουμε αυτήν την ε, υποχρέωση ως Προεδρία να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία μετά το Κοτονού. Ένα από τα σημαντικά σημεία στη συζήτηση αυτή είναι ότι φτάσαμε σε μια συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η συμφωνία μετά το Κοτονού θα πρέπει να προετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τις ατζέντα του 2030 των ΟΕΕ Εθνών για να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η συμφωνία μετά το Κοτονού. Να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι θα συνεχίσουμε εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε την εντολή διαπραγμάτευση του Συμβουλίου και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Οι προηγούμενε προεδρίες προσπάθησαν, δεν ήταν εύκολο. Εμείς θα την ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία πάντως στη δική μας προεδρία Έξι γύρι διαπραγματεύσεων. Είμαστε κοντά πλέον, πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ζέλε από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου κύριε Υπουργέ ε, που είστε εδώ για να γίνει αυτή η συζήτηση ε, για τους στόχους ε, της Προεδρίας σας και στον τομέα της πολιτικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ την κυβέρνησή σας. Είναι η πρώτη φορά που μια χώρα ε, οργανώνει μια συνεδρία σε Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ ενώ έχει και την Προεδρία της Ένωσης. Ε, σας ευχαριστούμε επίσης για τη συνέχεια που θα δώσετε στο Κοτονού δεν έχουν όλοι πάντα την ίδια στάση ώρες οι χώρες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν που δεσμεύεστε προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα από εκεί πέρα βεβαίως πιέζει ο χρόνος. Το 2020 ε, λίγη η διάρκεια της Συμφωνίας του Κοτονού και ελπίζω στην ε, διαπραγμάτευση να φτάσουμε σε μια οικονομική συμφωνία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση αυτά που συμβαίνουν στα που ισχύουν στα πλαίσια της Συμφωνίας του Κοτονού, ε, κάποιοι από τους Αφρικανούς εταίρους μας δεν ήταν ε, διατεθειμένοι στα πλαίσια της Οικονομικής Συμφωνίας να εγκρίνουν κάποιες παραγράφους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα πλαίσια όμως της Συμφωνίας Κοτονού το έκαναν αυτό. Αν λοιπόν δεν υπάρξει μια διάδοχος ε, συμφωνία που είναι και ίσως αυτό ένα ενδεχόμενο, τι θα γίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, μπορεί να πέσουμε στο κενό. Ένα αυτό. Δεύτερο, ε, μια παλαιά απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, την Συμφωνία του Κοτονού και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη ε, που συνδέονται αυτά τα δύο. Έχουμε τον προπολογισμό. η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Θέλουν να πάψει να ισχύει όμως η κάποια κρατημέλη από ό,τι ακούμε. Σε ό,τι αφορά τα νοσιωτικά κράτη, γίνεται λόγος για την κλιματική αλλαγή, αλλά ακριβώς ε, νησιωτικά και βόρεια κράτη φοβούνται μήπως ε, η ε, συνεργασία ε, όπως αυτή τη στιγμή ε, γίνεται μεταξύ ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρει ένα περιφερειακό χαρακτήρα ε, και μήπως υπάρξει υπερβολική εστίαση στην περιφερειοποίηση, περιφερειακή διάσταση υπέρ της Αφρικής. Και μείνουν εκτός άλλες περιοχές του κόσμου. Θα ήθελα λοιπόν στο πλαίσιο της δικής σας προεδρίας έχετε τώρα τη δυνατότητα, ε, είναι δυνατή μήνες για σας, να προωθήσετε αυτό το θέμα. Πρώτον, να φροντίσετε να μπει στο κενό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που είχαμε μέχρι τώρα στο ΕΤΑ, στο Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Ανάπτυξης, ε, να μην πάψουν να υπόκεινται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και εφόσον μπει ε, το ΕΤΑ στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, θα πρέπει να παραμείνει η συνεργασία υπό τη μορφή που έχει. Θέλω να υπάρξει αυτό το λεγόμενο ring fencing που λένε και οι Άγγλοι. Ευχαριστώ. Πήγατε κάπως πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ξέρω ότι ο ασχολείται και με αυτά. Ο οπότε γνωρίζει τα θέματα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Ζέλερ. Εκτιμώ το γεγονός ότι θέσατε αυτό το ζήτημα. Είχα μια συζήτηση χθες το απόγευμα με τον εκπρόσωπο εκπρόσωπο του Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι φορά την εισαγωγή στον προπολογισμό ούτως ή άλλως το θέμα θα έρθει στο, στο Κοινοβούλιο δεν θα χρηματοδοτηθεί πλέον από διάφορα ε, σημεία, διάφορες γραμμές των δαπανών όπως ισχύει ως τώρα ε, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε και να προωθήσουμε αυτή την ιδέα εμείς θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη συνένεση για το πολυμερές πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αριστερά της Προεδρίας μας ε, δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί βέβαια είναι μάλλον αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο λαμβάνοντα υπόψη το γεγονός ότι θα έχουμε τρεις μήνες ουσιαστικά τρεις ή μισή μήνες ε, πραγματική ουσιαστική δουλειά, γιατί έρχονται οι ευρωεκλογέ μετά. Αυτό που θέλουμε είναι όμω να θεσπίσουμε κάποιε προτεραιότητε, να έχουμε κάποιε γενικέ ιδέε ε, για το μελλοντικό προπολογισμό τη Ένωση. Και η δεύτερη προσέγγιση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να εγκριθεί αυτό στο το τέλος του 2019, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο εξάμεινο. Δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς. Εγώ συζήτησα πάντως με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν και ενδιαφέρονται ε, να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα της χρηματοδότησης ε, των χωρών ΑΚΕ. Θα βασιστούμε στην εντολή ε, του Συμβουλίου βέβαια για το θέμα αυτό και θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε όσο γίνεται περισσότερο την διαπραγμάτευση με τους συναδέλφους από τις χώρες ΑΚΕ. Όπως σας είπα, είναι προτεραιότητά μας για αυτήν την περίοδο. Βεβαίως, είπαμε, είναι 3,5 μήνες. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να φτάσουμε σε μία λύση. Γνωρίζω βεβαίως ότι είναι πολλές οι χώρες που ε, συνδέονται και διμερώς με κάποιες σημαντικές χώρες της Ένωσης. Υπάρχουν διάφοροι διάβλοι. Χρειάζεται όμως ένα σαφές πλαίσιο για τη χρηματοδότηση αυτής της συμφωνίας με τις χώρες ΑΚΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα συναντήσετε και την Αφρικανική Ένωση, όπως ξέρω, κύριε Υπουργέ, ε, διότι έχουμε δημιουργήσει και μια επιτροπή παρακολούθησης ε, από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να παρακολουθούμε ε, τη Συμφωνία του και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Είμαστε σε επαφή και με την Επίτροπο Νίμιτς που ασχολείται σχετικά. Και αυτό που ρωτήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι το εξή. Υπάρχει μια έλλειψη σαφήνεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία έχουμε την στρατηγία την Αφρική, από την άλλη έχουμε τη στρατηγία τη χώρα ΑΚΕ. Η στρατηγία την Αφρική αφορά το σύνολο τη Αφρική, αφορά και την Βόρεια Αφρική δηλαδή, που όμω εμπίπτει και στην πολιτική γειτονία. Πολλοί λοιπόν μα ζητούν, μα ρωτούν ε, πώ όλα αυτά συνδυάζονται. Καλό θα είναι αυτό σε πολιτικό επίπεδο στο μέλλον να διευκρινιστεί, διότι η εταίροι μα, η Αφρικανική Ένωση, θέλει να μιλήσει μαζί μας ως μία ενιαία οντότητα. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας διάλογος ε, για όλα αυτά τα ζητήματα εν εξελίξη. Επίσης οι χώρες της έχουν την αίσθηση ότι έχουν παραμεληθεί κάπως σε μια εποχή που χρειάζονται τη βοήθειά μας ε, λόγω των ζητημάτων που προκύπτουν με την κλιματική αλλαγή. Ε, στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο Παρίσι είναι συμμαχοί μας ε, και σε άλλα διεθνή φόρα. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε λοιπόν τον ειρηνικό και την ε, Καραϊβική. Δεν ξέρω αν θέλουν να θέσουν άλλες, άλλες ερωτήσεις συνάδελφοι. Ιδάλλως ε, κάτι ακόμα θέλω να πω, κάτι πρακτικό. Αν το έχετε υπόψη. Το ελληνικό συνέδριο έκανε μια έκθεση για τη ΜΚΟ στον ανθρωπιστικό τομέα και το πώς ε, επιχειρούν επί τόπου. Είχαμε μια συνάντηση με κάποιους ΜΚΟ πριν τα Χριστούγεννα. Υπάρχει... Υπάρχουν οι μεγάλες ε, ΜΚΟ, οποίες χρησιμοποιούν τοπικές NGOs, ΜΚΟ για την υλοποίηση των πολιτικών. Και εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα διαφάνεια, πώ μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, λέει το Συνέδριο, ότι η χρηματοδότηση πάει στους κατάλληλου ανθρώπους. Ε, Η ΜΚΟ όμως ε, θα πρέπει να λάβουν, να λάβουν υπόψη πόσο δύσκολο είναι να επιχειρήσουν σε κάποιες χώρες. Όταν δίνουμε κάποια ενίσχυση ε, σε, ε, σε Σύριους πρόσφυγες εντός της Συρίας, δεν μπορούν να πάνε εκεί οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τοπικές ΜΚΟ. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό, το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους. Η άλλη δυσκολία την οποία εγώ δεν γνώριζα ήταν και ο Ενρίκη και όταν συζητήσαμε με τον Ρόι. ε, υπάρχουν και η νομοθεσία, υπάρχει νομοθεσία κατά τη τρομοκρατίας και ειδικά του ξεπλήματο χρήματο που επηρεάζει την ανθρωπιστική δράση επιτόπου. Ε, κάποιες τράπεζες είναι επιφυλακτικέ στο να μεταφέρουν χρήματα από την Ευρώπη ε, προς χώρες όπως το Νότιο Σουδάν ε, ή τη Συρία. Αυτό σημαίνει όμω ότι ε, αυτοί που εργάζονται στην ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχουν μαζί τους ε, χρήματα σε ρευστό, δεκάδες χιλιάδες ε, δολάρια ε, και βεβαίως αυτό γνωστοποιείται και μετά αποτελούν στόχο. Ορισμένε καλέ προθέσει λοιπόν σε κάποια νομοθεσία να σταματήσει και το ξύλιμα χρήματο, παραδείγματο χάρη, είναι ορισμένε φορέ έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Κάποιοι υπουργοί το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το Συμβούλιο το έχει συζητήσει. Θα πρέπει πάντω να εξασφαλίσουμε ότι το τραπεζικό μα σύστημα θα αντιληφθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται υπό δύσκολε συνθήκε στον ανθρωπιστικό τομέα και πρέπει να μην περιπλέξουν ακόμα περισσότερο το έργο του ε, σε πρακτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Δεν ισχύει αυτό για αυτούς που δουλεύουν στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στη Συρία και στην Εμένη και σε άλλα μέρη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα δεν λειτουργεί ε, η μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών. Όλοι προσπαθούν ε, να ε, προσπαθήσουν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ανάγκες. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ΚΟΑΤΟ και η ΚΟΝΤΕΦ, δύο πολύ σημαντικές ε, οργανώσεις, είχαν ε, ε, συζήτηση κοινή την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο και προετοιμαζόμαστε με το Συμβούλιο για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να χρηματοδοτούν την αρρωγή που παρέχουν. Γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες ε, λειτουργούν, δρούν επί τόπου και θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να διευκολυνθεί η εργασία τους. Χαίρομαι, χαίρομαι που έφτασε το θέμα στις επιτροπές ε, του Συμβουλίου, γιατί άκουγα ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα ρωτήσουμε βέβαια και τον Επίτροπο Στυλιανίδη το απόγευμα. Ωραία. Ε, μπορούμε να σας ελευθερώσουμε αν δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις. Ε, μία και τριάντα έχουμε και γεύμα με τους συντονιστές. Ευχαριστούμε που ήρθατε και σας εύχομαι τα καλύτερα.